Τώρα, για την υπογραφή των ε, πράξεων που έχουν ε, υιοθετηθεί υπό την κανονική νομοθετική διαδικασία θα υπογράψουμε το, μαζί με το Συμβούλιο σύμφωνα με τον κανονισμό 74 του κανονισμού του Κοινοβουλίου τα, όσα εγκρίθηκαν στην προηγούμενη σύνοδο ε, και θα είναι διαθέσιμα για όλους σας από το